Okay. Philip. We start. Καλημέρα. So, listen now. I will speak Swedish. Uh, Två meddelanden. Θέλω να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Uh, Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάτι εκτός ε, θέματος και εκτός ημερησίας διατάξεως. Θεωρείτε τον εαυτό σας υποχρεωμένο να απαντά στα γράμματα των μελών της Επιτροπής Απασχόλησης, ναι ή όχι. Γιατί σας έχω στείλει επανειλημμένως για διάφορα θέματα γράμματα και δεν έχω λάβει απάντηση. Και η τελευταία απάντηση που θα ήθελα να μου στείλετε είναι πώς εξηγείτε το ότι στην, ε, ε, ψηφίζοντας για την οδηγία για το χρόνο εργασίας στις οδικές μεταφορές βρέθηκε να υπάρχει μία ψήφος παραπάνω από τα παρόντα μέλη στην ψηφοφορία. Δεν έλαβα την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ο γραμματέας μου λέει ότι δεν έχει δει τις επιστολές, δεν ξέρω. Αν, αν το έχετε στείλει στη γραμματεία θα το εξακριβώσουμε και μετά θα σας ε, δώσω την απάντηση. Δύο ανακοινώσεις θα κάνω τώρα. Πρώτον, για την κινητικότητα των ασθενών και τη σχετική οδηγία. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Εγώ και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς Επικαλούμαστε το άρθρο 47 για ενισχυμένη συνεργασία και άρα προτείνουμε η καθήλια αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, να μην ψηφίσει για την παράγραφο 69. Είχαμε συνάντηση με τον κύριο Καλαιότα και τον κύριο Πέτεριν και τους τρεις προέδρους την περασμένη εβδομάδα. Αλλά υπάρχει ο κανόνας 47, όπως σας είπα, που λέει ότι τελικά ο πρόεδρος της ε, ε, καθήλης αρμόδιας επιτροπής αποφασίζει ε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν ήθελε να ακολουθήσει αυτόν τον κανόνα 47, ο πρόεδρός της δηλαδή, και θέλει να ψηφίσει και τις δικές μας τροπολογίες. Παρόλα αυτά καταλήξαμε σε κάποιο είδους συμβιβασμό, ότι δηλαδή θα δώσουμε την ευκαιρία στη δική μας Επιτροπή να υποβάλουμε εκ παραλίλου στην Ολομέλεια ε, τα, τις δικές μας τροπολογίες με 40 βουλευτές. Ο κύριος Σίσκου μας είπε ότι πρόκειται για έξι από τις δικές μας τροπολογίες ε, οι οποίες τελικά δεν θα ε, ψηφιστούν. Οι υπόλοιπες θα ψηφιστούν. Ο γραμματέας θα εξετάσει την κατάσταση για να δούμε αν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, και θα επανέλθουμε και θα συγκεντρώσουμε 40 βουλευτές. Ε, θα είμαστε σε επαφή με τον κύριο Μπραγκέ, το πήγαμε μαζί στη συνεδρίαση και επί τη βάση αυτού, ξαναλέω, εκ παραλίλου θα υποβάλουμε τις δικές μας τροπολογίες αν θεωρούμε ότι η στάση που θα τηρήσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος αποκλίνει πάρα πολύ από τη δική μας σήμερα ψηφίζουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα γίνει αυτή η ανάλυση από τη γραμματεία που σας έλεγα και θα επανέλθουμε. Αλλά θέλουμε να προσυπογράψετε φυσικά τις δικές μας τροπολογίες και θα τις υποβάλουμε εκ παραλίλου. Αρχίζουμε με την έκθεση της κυρίας Λάμπερτ Στη συνέχεια το, την έκθεση του κυρίου Γιάνν Κράμερς και μετά τη δεύτερη της κυρίας Λάμπερτ αλλά και μετά θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ψηφοφορίες αλλά σας τα είχα πει ήδη αυτά. Λοιπόν, αρχίζουμε με την έκθεση, την ομοδότηση της κυρίας ε, Λάμπερτ, συμβαστική α, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, καταπίπτει η δεύτερη τροπολογία της εισηγήτριας. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, καταπίπτουν ναι, οι 8, 7 και 9 και πάμε στη συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 10. Ε, ψηφίζουμε την 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 3 και 4 καταπίπτουν. Συμβαστική F ε. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν διάφορες τώρα και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε παρακαλώ. Άρχιδη ψηφοφορία. Yeah, yeah, I know. okay. Oh, two persons who don't have it. You're not fast enough, Harold. <laughs> yeah, put it in. So, omröstningen avslutad. Πέρας. εψήφισαν, ε, οι 33 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Ε, συγχαρητήρια κυρία Λάμπερτ. Herr Γνωμοδότηση του, του κυρίου Κρέμερ. Κρέμερ για ε, όλα τα παραρτήματα. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. False. Yeah. No, no, we have to vote on the first part because the second part is, is, is withdrawn. Okay. Okay. Φύγαν, θάλο. Τέσσερα καταπίπτει. Οι δύο και τρία θεωρούνται και κρυμμένες. το, την ε, υπαριθμόν 1 πρέπει να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα για το δεύτερο ήρθηκε. Λοιπόν, η πρώτη τροπολογία υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Ε, ε, αλλά Ψηφίσατε όλοι. Όσοι δεν έχουν κάρτες πρέπει να μας πείτε πώς ψηφίσατε, να μας, ε, να μας ενημερώσετε. Κύριε Πινέντα, δύσκολο είναι, δεν μπορείτε με το μηχάνημα, δεν δουλεύει. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας,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 41 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν 43, 44 και 45 και ψηφίζουμε την 46 υπέρ. Κατά. Ισοψηφία μάλλον. 46 ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε ηλεκτρονικά για την 46. Ε, να ήρθω. Ε, Όμως είναι Πέρας ψηφοφορίες 38 ψήφισαν. 18 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ και 54 μαζί κατά αποχές εγκρίνεται 51 καταπίπτει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 Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Θέλει ηλεκτρονική εξακρίβωση για την 67. 67 ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρασε. 19 προς 19 ισοψηφία. Ε, άρα απορρίπτεται. Λόγω ισοψηφίας 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ 72 κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76, ε, 77 και 78 καταπίπτουν και ψηφίσουμε την 79 υπέρ. 79 υπέρ. Κατά. εκεί εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. εκεί εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. εκεί εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. εκεί εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και καταπίπτουν διάφορες τροπολογίες μέχρι την 87. Ψηφίζουμε 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική D. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται κατά καταπίπτουν 92 και 94 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 με προφορική τροπολογία προσθέτουμε, ε, διαγράφουμε το end sheltered employment υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 82 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στα εκτιμώντας 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 ε, υπέρ κατά Ε, και πάλι ψηφίστε για την 20 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, όχι, ηλεκτρονικά λοιπόν πάλι για την 20 γιατί δεν ξέρω. Ηλεκτρονικά ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 41 ψήφισαν, ε, ε, 21 ψήφι προς 19 εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε και αυτά. Okay. Τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τρία υπέρ. Μπορούμε αν μπλοκ να τα ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε. Αλλά Ρωστάτ. Ψήφισαν όλοι. Αλλά Ρωστάτ. Ψηφίσατε. Omröstningen har ut... 42 ψήφισαν 25 υπέρ, 2 κατά και 15 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Λάμπερτ. Πάμε στην έκθεση του κυρίου Πινέιντα για την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα. Don't know your page. I have my page. Δεν ξέρω εσείς τι έγραφα, έχετε και σε ποια σελίδα είστε εσείς. Ξέρω που είμαι εγώ. Okay. Okay. Okay. 62 an Eurostar. 62 αρχίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 καταπίπτει. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. What is it? Εκτός μικροφώνου κυρία Μαντέιρα. Some internal problems. We go on 65 ε, υπέρ. Το δεύτερο τμήμα αποσύρεται. Για το πρώτο ψηφίστε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τρία της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά Εποχέ. απορρίπτεται 19 τη Επιτροπή Γυναικών υπέρ κατά Εποχέ. γκριντ 67 αποσύρεται 69 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 68 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται Συμβαστική α, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έκον 2 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το εξακριβώσουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική C. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αλλά Ψηφίσατε όλοι πέρα. 21 ψήφοι υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. 80 δεν καταπίπτουνε, 82 τώρα υπέρ. Ναι, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι δύο της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκον 7 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 6 και 8 καταπίπτουν 2 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MV3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. MV6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 20 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 86, 87 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι δύο της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ Δεν είναι ξεκάθαρο. Ηλεκτρονικά. Πρέπει να ψηφίσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Αλλά Ψήφισαν όλοι 22 υπέρ, 18 ε, κατά εγκρίνεται. Ε, συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Where were I? 113. 113. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 προφορική, ναι. 120 ψηφίσματα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική M υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, καταπίπτουν διάφορες τώρα, ε, μάλλον οι επόμενε επιτροπές γυναικών και φτάνουμε συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 140 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές επίσης εγκρίνεται. 149 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 συγγνώμη υπέρ. Ναι κύριε Μπιούσελ Μάθιος, συγγνώμη, ε, κάτι μικρό, μόνο γλωσσικό για την 149 το περάστε δεν επηρεάζει την ψηφοφορία, λέμε στα αγγλικά... Ε, μιλάμε για το οικονομικό καθεστώς, economical status. Είναι λάθος τα αγγλικά, economic status πρέπει να πούμε. Τέλος πάντων δεν νομίζω να δημιουργεί αυτό πρόβλημα σε άλλες γλώσσες. Καλά σας ευχαριστούμε. 150 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 147 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 151 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 152, μόνο το πρώτο τμήμα, το δεύτερο αποσύρθηκε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχέ Απορρίπτεται. 155 μόνο το πρώτο τμήμα γιατί το δεύτερο το έχουμε αποσύρει υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 164 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ψηφίστε κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική ε, ε, μικρόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πι υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 αποσύρεται 177 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται 178 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 179 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ. Κατά Αποχέ, εγκρίνεται 181 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 183. 183. Την 182 την ψηφίσαμε αφού εγκρίθηκε. Ο καλά. Να το εξακριβώσουμε. Ψηφίστε ηλεκτρονικά για την 182. Όμως δεν είναι Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 24 προς 15. Εγκρίνεται. 183 τώρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική Q υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. «187 σας λέω». Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188 αποσύρεται. 189 τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 τώρα κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 196 καταπίπτει. 195 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Α, αποχές απορρίπτεται. Η υπαριθμόν 1 ε, υπέρ. Τη ζητήσεων ομάδων unblock. Όλες μαζί. Ψηφίστε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα στα σε συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και καταπίπτουν διάφορες τροπολογίες και φτάνουμε στη συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, η 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ. Κατά απο... αποχές απορρίπτεται. MVC της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά, εξακρίβως παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Αλλά ώστε... Ψήφισαν όλοι. 22 ε, προς 18 εγκρίνεται 38 υπέρ 37 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά Αποχές. Ο κύριος Λιντέ. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Έγινε... Υπάρχει ένα λάθος στη μετάφραση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ψηφίσουμε το 37 και όχι 38. Μπορείτε να ξαναρχίσουμε, μπορούμε να ξαναρχίσουμε την ψηφοφορή. Ναι, ήταν η 37. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτευ. Συμβαστική 7. Ε, ε, ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η δίτη της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτε 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51-52 αποσύρονται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ 59, ε, κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ωραία ψηφίστε παρακαλώ Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 40 ψήφισαν. 38 υπέρ. 2 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Πινέδα. Ο ε, κύριος Μπουσιλ Ευχαριστώ ε, πολύ. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε συζητώντας με το Steven Χιούς αντιλαμβάνομαι ότι κανονικά η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί χωρίς συζήτηση ή στην Ολομέλεια. Είναι ένα πολύ βασικό θέμα και ε, δεν πρέπει να περάσει έτσι αθόρυβα. Εάν όμως ε, συμφωνήσουμε όλοι μπορούμε να ζητήσουμε ε, να γίνει κάποια συζήτηση επί του θέματος. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε ε, είναι θέμα αποφάσεως για τις πολιτικές ομάδες. Θα συζητηθεί στις πολιτικές ομάδες και εγώ θα στηρίξω τη θέση σας. Προχωράμε. Στην έκθεση της κυρίας Τάουνερ για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η 8 αποσύρεται. 39 υπέρ κατά ε, αποχές απορρίπτεται 37 αποσύρεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 9 αποσύρεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται ένα υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται η 11 αποσύρεται 42 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται η 12 γλωσσικό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 αποσύρεται 2 της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14-15 αποσύρονται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 αποσύρεται 18 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20-21 αποσύρονται 43 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 αποσύρεται 23 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 αποσύρεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 αποσύρεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 αποσύρεται 4 της Επιτροπή ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 αποσύρεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 1 αποσύρεται, ε, η 1 ρέτζι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 και 3 αποσύρονται 4 και 35 ταυτόσημες μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 5 αποσύρεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οι 6 και 7 αποσύρονται πάμε στην τελική ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι πέρας. 23 ε, ε, υπέρ, 11 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Στην, ε, σε όλη την Επιτροπή. Κυρία Στάουνερ, πρέπει να κάνουμε τριμερή... Τώρα πρέπει να γίνει μια, ένας τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και εφόσον καταψηφίσατε θα πρέπει να παρουσιάσετε στον τριμερή διάλογο τη θέση ε, της Επιτροπής εγώ δεν έχω πρόβλημα εάν ε, το δεχθείτε, αλλά πρέπει να υπεραμεινθείτε τις θέσεις της Επιτροπής. Διότι διαφορετικά εγώ ο, σαν πρόεδρος μπορώ να παραστώ. Ευχαριστώ για ε, ε, καταρχήν για τη μεγαλοψυχία σας γιατί ε, με συγχαρήκατε μετά ευχαριστώ για τα μαθήματα βεβαίως δεν χρειάζομαι μαθήματα ξέρω τι θα κάνω είναι προφανές Είμαι, είμαι σοβαρός όμως. Από εσά εξαρτάται. Εάν δεν συμφωνήσετε με τη θέση μας, εγώ μπορώ να το αντιληφθώ και το σέβομαι. Αλλά στον τριμερή διάλογο θα πρέπει να ε, υπεραμεινθείτε τις θέσεις της Επιτροπής. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Μπορείτε να το σκεφτείτε αν θέλετε. Πάμε στην έκθεση της κυρίας Μαντέιρα για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας για τις εγγύους και τις λεχόνες. Κύριε Μαντέρα, έχετε στήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να σας ενημερώσω ότι η τροπολογία 40 έχει και μια προφορική τροπολογία μαζί της κυρία Στάουνερ. Αυτά ήθελα να σας πω. 40, ναι, ωραία. Α, και η κυρία Σρόντερ. Κυρία Σρόντερ, διαδικαστικό. Oh, zum... Ακριβώς, σχετικά με την τροπολογία 21, 21 αλλά ποιος ε, είναι στον κατάλογο σχετικά με την ε, ε, τροπολογία αυτή η οποία περιλαμβάνεται και είναι σημειωμένη στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ωραία, θα ψηφίσουμε τώρα. 22 υπέρ. Κάταμα. αποχές συγκρίνεται. 23 υπέρ.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 κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 αποσύρεται 40 υπέρ Α, έχουμε και την προφορική τροπολογία που μας λέγεται κυρία Στάουνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το 40 συμφώνησα με την εισηγήτρια γιατί το συζητήσαμε εχθές πρόκειται για την κατανομή των εβδομάδων πριν και μετά τη γέννα εγώ λοιπόν ε, θα πρότεινα να ε, ψηφίσουμε το κείμενο για έξι εβδομάδες πριν από τον τοκετό έτσι το έχουμε συμφωνήσει, τελεία εκεί και το υπόλοιπο θα διαγραφεί. Ευχαριστώ. Ωραία, κυρία Μαντέρα, το, σκεφ... το δέχεστε. Ε, μπορεί να το επιβεβαιώσει η κυρία Στάουνερ αν θέλει. Αποσύρουμε όλο το τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή έξι εβδομάδες πριν από τη γέννηση και μετά εντάσσεται το υπόλοιπο στην τροπολογία. Άρα φτάσαμε υπέρ της πρότασης. Ωραία, με αυτή την προφορική τροπολογία ψηφίζουμε τη 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 42. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 και 49 είναι ταυτόσιμες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική B υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 12 ε, και 53 καταπέπτουν 13 ψηφίσματα υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Οι φιλελεύθεροι τι κάνουν. Γιατί 13. 13, 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 4 ναι. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 16 και 17 αποσύρονται. 18 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21 με προφορική τροπολογία ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κύριε Μαντήρα ε, Η προφορική αυτή τροπολογία σημαίνει υπερψήφιση της 21. Δηλαδή, εάν δεν αποσυρθεί αυτή η, φράση, τότε θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε. Νομίζω ότι έγινε ένα λάθος στην ψηφοφορία. Είπα με την προφορική τροπολογία. Το είπα με την προφορική. Ψηφίζουμε την 21 λοιπόν υπέρα. Κατά. Εποχέ συγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψήφιζαν όλοι. Πέρασε. 29 υπέρ, 3 κατά μία αποχή. Γκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μαντέιρα. He woke up when he heard the word. now we have three things. Three things. Yeah? Okej. Nu har vi Ωραία, πάμε στη σύμβαση του ΟΗΕ τώρα. Της κυρίας Γέλαβα. Έχουν αποσυρθεί ε, διάφορες τροπολογίες. Ψηφίζουμε την ε, νομοθετική πρόταση μόνο, ηλεκτρονικά, την νομοθετική πρόταση μόνο. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. 33 υπέρ, κανένας κατά, μια αποχή. Συγχαρητήρια, κυρία Γελέβα. Το ίδιο και για το πρωτόκολλο. Για την νομοθετική πρόταση ψηφίζουμε μόνο. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. 34 υπέρ μία κατά, καμία αποχή. Και πάμε στο ψήφισμα τώρα. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4. Με προφορική τροπολογία. Ε, την ημερομηνία αλλάζουμε δηλαδή υπέρ. Πρέπει να ξυπνήσετε τώρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για την παράγραφο 7. Είχαμε μια προφορική τροπολογία και έχετε το κείμενο. Για την παράγραφο 7 ψηφίζουμε. Παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά, κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Citation 9β με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα δηλαδή. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 33 ψήφισαν. 32 ε, υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Γέλεβα. Πέρας των ψηφοφορίων. Φίλιπ. Εντάχει θα ήθελα να πω ότι σε δύο εβδομάδες ε, θα γίνει μια συνεδρίαση. Νομίζω, εγώ δεν μπορώ να παρευρεθώ και νομίζω και οι συνάδελφοι θα μπορέσουν. Αυτή είναι η τελευταία μου συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τους συναδέλφους για τη βοήθειά τους και για την εξαιρετική συνεργασία, την αγαστή αυτή συνεργασία και σας ευχαριστώ που μερικές φορές συμφωνήσατε μαζί μου. Σας ευχαριστώ όμως γιατί πάντα με ακούγατε είτε συμφωνούσατε είτε όχι. Και εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω. Εγώ θα είμαι εδώ στις 16, τότε θα είναι η τελευταία μου συνεδρίαση σε αυτή την Επιτροπή και Φυσικά δεν συμφωνούσαμε πάντα σε πολιτικά ζητήματα, αλλά είχαμε πολύ ανοιχτές σχέσεις και πρέπει να σας ευχαριστήσω και εγώ γιατί μας βοηθήσατε ιδιαίτερα. Ήσασταν πάντα ευδιάθετος και είχατε συνεισφέρει για την καλή διάθεση αυτής της ε, συνεδρίασης. Στίβεν, και εγώ δεν θα είμαι εδώ στις 16, ε, γι' αυτό θα ήθελα να απηχήσω τα όσα ελέγχθηκα με την εξαίρεση ότι σας ευχαριστώ γιατί συνήθως συμφωνούσατε μαζί, μαζί μου. Χαίρομαι για τα δέκα χρόνια συνεργασίας με τα πάνω και τα κάτω τους και θα ήθελα να ευχαριστώ στον κύριο Μπούσχιλ Μάθιους καλή συνταξιοδότηση. Ο Στίβεν σίγουρα, σίγουρα θα, θα του λείψει του Στίβεν. Ωραία. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το Ταμείο για την Αντιμετώπιση της Παγκοσμιοποίησης, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Αφορά λοιπόν το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και εδώ υπάρχει ένα αίτημα από μια ισπανική εταιρεία, από μια ισπανική Καστίγια Ηλεών, η Αραγών. Άρα θα ψηφίσουμε στις 16. Ε, η κυρία Στάουνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Πρόκειται όπως είπαμε για μία αίτηση της Ισπανικής κυβερνήσεως της Καστήλης Λεών και Αραγκών και υπάρχει και μία αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τεχνική βοήθεια. Είναι δύο θέματα που μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε μαζί και έχει ήδη γίνει μία συζήτηση με τους κοιόδης εισηγητές όπου έχουν διατυπωθεί ορισμένα ερωτήματα και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί τώρα να μας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να προσθέσω κάτι καινούριο και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας πει τι μέλη με την τεχνική βοήθεια και ε, εάν ε, είναι ήδη ε, εδώ μπορεί να μας πούν για τις ερωτήσεις που έχουμε θέσει στην Ισπανική κυβέρνηση σχετικά με την ενίσχυση της ε, βιομηχανίας ε, ε, παραδόσεως των αυτοκινήτων και είναι μια αίτηση η οποία είχε υποβληθεί το Δεκέμβριο και ανανεώθηκε το Φεβρουάριο διότι τότε ήταν δυνατή να υπάρχει συγχρηματοδότηση της Ισπανικής ε, κυβερνήσεως η οποία δεν προϋπήρχε και γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω αν στο τελευταίο δεκαπενθήμερο έχει προκύψει κάτι καινούριο και περιμένω μία ενημέρωση. Ευχαριστώ. Ε, λέω να προχωρήσουμε όπως ε, πρότεινε η κυρία Στάουνερ πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν οι απαντήσεις ε, και μετά θα δώσω το λόγο στην Ισπανική κυβέρνηση αλλά καταρχήν η Επιτροπή Ευχαριστώ η κατάσταση έχει ως εξής ο ε, κανονισμός προβλέπει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι 0,35% των 500 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνική ενίσχυση. Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνει μια τέτοια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο λόγος είναι ότι έχουμε χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις μας για να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε αυτές τις, ε, ε, τις αιτήσει για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε όσο το δυνατόν πιο, πιο γρήγορα αυτούς που χρειάζονται αυτή την ενίσχυση. Για το 2009 τίνουμε 500 ε, εκατομμύρια ευρώ διότι χρειάζεται να ξεκινήσουν ε, δραστηριότητες που δεν μπορούσαν να ε, χρηματοδοτηθούν διαφορετικά. Πρόκειται για τα εξής. Καταρχήν πληροφόρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να καταρτήσει μία ιστοσελίδα σχετικά με αυτό αυτή την ε, εργασία ενισχύσεως και το έχουμε πρέπει να, να συνεχίσει και την εργασία της. Δηλαδή η ισοσελίδα αυτή είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους. Επίσης θα θέλαμε να τυπώσουμε αφίσες για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε ε, την ενημέρωση σχετικά με αυτό το Ταμείο Προσαρμογής και συγχρόνως να αναλάβουμε διάφορες ε, ε, δημόσιες σχέσεις ε, σχετικά με την ηλεκτρονική μετάδοση. Έχουμε μία συνεδρίαση με τις εμπειρογνώμονες. Έχουμε ήδη ε, οργανώσει δύο ε, δύο συναντήσεις και ελπίζουμε ότι μέσα στο 2009 θα έχουμε δύο ακόμη συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονες αυτούς για να εξετάσουμε το νέο κανονισμό και να βεβαιωθούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν αντιληφθεί τις δυνατότητες του Ταμείου αυτού προσαρμογής. Συγχρόνως θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση. Πρέπει από τώρα να ξεκινήσουμε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ε, ε, στη μέση της διαδρομής ε, την εφαρμογή του κανονισμού γι' αυτό και ξεκινήσαμε το 2009 για να προλάβουμε να ετοιμαστούμε. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να ετοιμάζουμε την παρακολούθηση και τον έλεγχο αλλά ε, όπως σας είπα δεν μπορούμε να ζητήσουμε άλλες ε, πιστώσεις για το 2009 διότι έχουμε ε, προσφέρει όλες τις ε, αναγκαίες πληροφορίες εις ε, τις δημοσιονομικές αρχές. Η πρότασή μας είναι μικρότερη από το ανώτατο δυνατό επίπεδο αλλά αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα. Θέλετε να αναφερθώ τώρα στην ισπανική περίπτωση. Εντάξει, σχετικά με την περίπτωση αυτή πρόκειται για μία πρόταση η οποία μοιάζει με άλλες προτάσεις τις οποίες έχετε ήδη συζητήσει δηλαδή για 1082 πωλήσει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση της αγοράς αυτοκινήτων και της βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και διαπιστώνουμε ότι μειώνονται οι συμμετοχές μας στις τρίτες αγορές, στις αγορές των τρίτων χωρών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η ε, κατάσταση της βιομηχανίας στην Ισπανία επιβεβαιώνεται από τις στατιστικές. Δηλαδή, Πρόκειται, ε, ε, εάν ο αριθμός αυτός των απολύσεων είναι σωστός, πρόκειται για 1080 απολύσεις στα πλαίσια 12 επιχειρήσεων για τα πλαίσια της ε, δράσης ΝΑΣ 2 για την ε, κατασκευή αυτοκινήτων και κινητήρων αυτοκινήτων ε, έχουν σεβαστεί το νεάμινο που επιβάλλεται και γι' αυτό το λόγο είμαστε ε, έτοιμοι να αποδεχθούμε την αίτηση και ε, διότι θεωρούμε ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις. Όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες για τα άτομα τα οποία πρόκειται να απολυθούν πρόκειται για ένα σύνολο μέτρων που αναφέρεται σε ένα αναπροσανατολισμό των ατόμων αυτών για να μπορέσουν να βρουν μια άλλη θέση εργασίας Πρόκειται για 350 άτομα τα οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν συγκεκριμένα και η κατάρτιση αυτή προτείνεται βάσει των συμφερόντων τα οποία, των ενδιαφερόντων που έχουν εκφράσει οι απολυμμένοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Θα ε, υπάρξει ε, υλικό ε, ηλεκτρονικό ε, θα βελτιώσουν τις δεξιότητες που έχουν ήδη δηλαδή αυτοί που εργάζονται σε αποθήκες μπορούν να διαχειριστούν την ε, διοικητική μέρημνα και ούτω καθεξής πρόκειται για διάφορους συνεργάτες οι οποίοι χάρη στις γνώσεις τους θα μπορέσουν να ε, ε, να ξαναεργαστούν εάν ε, βελτιωθούν οι δεξιότητές τους και αυτό είναι δυνατόν μέσω των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων και τέλος πρέπει να υπάρξει επαγγελματική κατάρτιση για να μπορέσουν να υποφεληθούν και από άλλα μέτρα, δηλαδή τις δυνατότητες να βρουν ε, μία δουλειά, να ψάξουν για μία δουλειά ενεργά και υπάρχει ένα ποσό 300 ευρώ το μήνα που προβλέπεται να στηρίξει αυτές τις ε, εργασίες ε, εντάξεως στην αγορά εργασίας. Αυτή η υπόθεση δηλαδή μοιάζει πολύ με άλλες τις οποίες ήδη έχετε παρακολουθήσει και δεν υπάρχει τίποτα που να την καθιστά ιδιαίτερη. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δεχθείτε αυτή την ε, πρόταση. Ωραία. Εδώ μιλάμε για δύο θέματα, φενός για την τεχνική βοήθεια, ε, ιστοσελίδες και τα λοιπά, τα οποία προβλέπονται στο κανονισμό και υπάρχει ένα ανώτατο επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να πληροφορήσει και υπάρχει και η συγκεκριμένη περίπτωση της ε, ε, της ε, ε, Ισπανίας. Ο κύριος Πενέντα έχει το πρώτο στον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που προείπε η Επιτροπή και δέχομαι αυτή την υποστήριξη. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ήδη τάχθηκε υπέρ και νομίζω ότι είναι αποφασιστική σημασίας η παρέμβαση της, δηλαδή Θεωρώ ότι η Επιτροπή μας έχει αρμοδιότητες, αλλά τις βασικές αρμοδιότητες έχει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και γι' αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσουμε εδώ προβλήματα. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την χρηματοδότηση αυτή. Άρα νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να εγκριθεί εντάχει χωρίς αντιρρήσεις από τη δική μας πλευρά. Ο κύριος Εσκόβαρ, ευχαριστώ και εντάχει θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γκαμπριέλα Στάουνερ, διότι ξέρω ότι παρακολουθεί εκ του σύνεγγης αυτό το μέσον και εργάζεται επί του θέματος. Εγώ γνωρίζω την κατάσταση που ζει η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία που είναι τραγική για δύο λόγους. Διότι ε, ζούμε μία τραυματική στιγμή και αυτές οι μικρές επιχειρήσεις έκαναν μία σειρά επενδύσεων και τώρα με την πιστοτική αυτή ε, ξηρασία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην ε, αποπληρωμή των επενδύσεων η κατάσταση είναι δραματική. Πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι και οι μοναδικές μέσα στα πλαίσια του οικονομικού και κοινωνικού ιστού αυτών των περιφερειών. Εγώ διάβασα όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε η Επιτροπή και οι επιπρόσθετες πληροφορίες που μας έδωσαν οι Ισπανικές αρχές και επειδή δεν ε, υπάρχει αντίθετη γνώμη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, θα ήθελα να γίνει αυτή η μεταφορά. Και μέσω μίας επιστολής νομίζω ότι θα έπρεπε να εγκρίνουμε αυτό το θέμα της χρηματοδότησης εντάχει. Ευχαριστώ. Σημερίζομαι την άποψη του κυρίου Πενέντα και δέχομαι αυτά που προείπε. Okay, Η κυρία Στάουνερ για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ ε, για τα σχόλια. Δεν θέλω απλώς να σας πω ότι όσον αφορά την τεχνική βοήθεια για το 2009 ο συνάδελφος Ευρωπαϊκής Επιτροπής το γνωρίζει ήδη αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ε, να διατεθούν τα χρήματα όλα ε, προς όφελος των ε, εργαζομένων και όχι για προώθηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, αν χρηματοδοτείται μία ιστοσελίδα που ήδη υφίσταται όπως γράφει η Επιτροπή από το 2007 και το 2008 στις εκθέσεις της πώς συνυπολογίζεται το κόστος της τώρα καθώς και άλλες δαπάνες για ε, μία δημοσιοποίηση του Ταμείου δεδομένων των προτάσεων οι οποίες υπάρχουν δεν νομίζω ότι αν αυτά είναι δεν νομίζω ότι αυτά είναι απαραίτητα και σχετικά με την ισφανική περίπτωση πρέπει να δω ακριβώς τα στοιχεία διότι ε, η ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού έχει συνενέσει και συμμετέχει και ο κύριος Πενέδα θα τα δω αλλά η Επιτροπή Προϋπολογισμού αν κατάλαβα καλά δεν μπορεί να προεξοφλήσει και να δεχθεί αυτή την ε, ε, πρόταση εάν δεν το έχουμε ζητήσει καν γνωμοδότηση. Δηλαδή δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τις δυνατότητές μας και τις αρμοδιότητές μας. Έχω όμως ε, επιφυλάξεις για την τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο τρίτο έτος του, του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης όλες, ε, όλα τα προβλήματα δεν, έχει, δεν έχουν λυθεί αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε για τις επόμενες 15 μέρες μέχρι ότου συζητηθεί τελικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή μας Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πενέρα, ο κύριος Κοτινή και ο κύριος Εσκομπάρ όσον αφορά την ιστοσελίδα και άλλες ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια που προβλέπεται εις τον κανονισμό και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά είναι κάτω από το ανώτατο ε, δυνατό επίπεδο. Είναι καλό να έχουμε ε, πληροφορίες για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Θα ήταν παράλογο να μας δοθούν οι πληροφορίες αυτές. Και δεδομένη της εμπλοκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι πρέπει να συνενέσουμε. Όσον αφορά την ισπανική περίπτωση δεν έχουμε επισέλθει σε πολλέ λεπτομέρειε. Νομίζω όμως ότι είναι μέσα στα πλαίσια που προδιαγράφονται. Όντως η Επιτροπή Προπολογισμού το έχει συζητήσει αλλά δεν έχει καταλήξει ως συνήθως θα υπάρξει διάλογος και εγώ έρχομαι από μία χώρα όπου η αυτοκινητοβιομηχανία είναι βασικός τομέας και η χώρα μου δεν έχει ζητήσει ενίσχυση αλλά αντιλαμβάνουμε όμως τα προβλήματα της Ισπανίας. Υπάρχουν δυσκολίες με την αυτοκινητοβιομηχανία αυτή τη στιγμή και δεδομένης που κάναμε για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ε, μιλάμε για τους ανθρώπους που αισθάνονται αποκλεισμένοι, για τις απολύσεις. Πρέπει λοιπόν όταν αυτά συμβαίνουν να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε και αυτά που λέγονται είναι σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε θετικά στο θέμα αυτό αλλά η τελική μας απόφαση θα βγει στην επόμενη συνεδρίαση. Ήταν, ε, τέλος η συζήτηση αυτή. Ήταν η τελευταία το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η επόμενη συνεδρία είναι στις 16 του μηνός. Θα έχουμε τον ε, Επίτροπο Σπίτλα, αλλά η συνεδρία μας θα διαρκέσει μόνο το πρωί. Έχουμε τον κύριο Σπίτλα και άλλον ε, ένα προσκαλεσμένο και θα αποφασίσουμε σχετικά με το Ταμείο Πασγομιζιοποίησης ευχαριστώ για την προσοχή σας και λύεται η συνεδρία.